Good afternoon, colleagues. We will... Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Ξεκινάει η συνεδρίασή μας. there changes proposed on the agenda... Αν υπάρχουν αλλαγές για την ημερήσια διάταξη, δεν υπάρχουν μάλλον αλλαγές. Τώρα τα πρακτικά θα πρέπει να γίνουν δεκτά. Μέχρι τώρα δεν υπάρχουν σχόλια, συνεπώς θεωρούνται αποδεκτά τα πρακτικά των προηγούμενων συνεδριάσεων. Δεν έχω ανακοινώσεις. Το επόμενο θέμα, φορολογικές πολιτικές και ισότητα των φύλων. Οι εμπειρογνώμονές μας βρίσκονται εδώ. Στόχος της ακρόασης είναι να συζητήσουμε το πώς τα διαφορετικά φορολογικά συστήματα μπορούν να επηρεάσουν τα θέματα της ισότητας στα διάφορα κράτη-μέλη. Με χαρά καλωσορίζω σήμερα εμπειρογνώμονες που δέχτηκαν την πρότασή μας να πάρουν μέρος στην ακροασή και να παρουσιάσουν τις εμπειρίες τους. Εμείς προετοιμάζουμε μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας για αργότερα, σε μερικούς μήνες. Οι φορολογικοί νόμοι θεωρητικά είναι ε, ουδέτεροι σε φιλετικό επίπεδο, αλλά παρόλα αυτά δημιουργούν μερικές φορές για κοινωνικούς λόγους και για λόγους παράδοσης διαφοροποίησης. Θα δούμε λοιπόν πώς τα φορολογικά συστήματα αυξάνουν ή μειώνουν τη συμμετοχή των γυναικών, δίνουν κίνητρα στις γυναίκες να ασχολούνται με την επιχειρηματικότητα και αν βοηθούν να καταπολεμήσουν την ένδια. Είναι αρμοδιότητα φυσικά εν πολύ των κρατών μελών η συγκεκριμένη φορολογική πολιτική. Εμείς όμως οφείλουμε να εξετάσουμε την ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Θα ακούσουμε λοιπόν τις απόψεις των εμπειρογνωμόνων. Ελπίζω να έχουμε μια καρποφόρο συζήτηση. Θα δώσω το λόγο τώρα στους εμπειρογνώμονες μας. Η κυρία Κλάτσελ είναι από το Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Εθνών για την ισότητα των φύλων Ισλανδοί. Ασχολείται επίσης και με τον ακτιβισμό, τον φεμινισμό και είναι και σύμβουλος για θέματα ισότητας προϋπολογισμών, παγκοσμιοποίησης και γυναικείων οικονομικών. Θα σας δώσω το λόγο κυρία Κλάτσα. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι τιμή μου που είμαι ανάμεσά σας σήμερα. Πρώτη φορά ένα θεσμικό όργανο της Ένωσης ασχολείται ενεργά με το θέμα και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό και η αφετηρία για περαιτέρω έργα. Ιδιαίτερα αφού γνωρίζουμε ότι υπάρχουν σαφείς νομικές υποχρεώσεις που υποχρεώνουν τα θεσμικά όργανα και τα κράτη-μέλη να φροντίζουν για την ισότητα και να αποφεύγουν τις διακρίσεις και στη φορολογική πολιτική. Δεν θα υπησέλθω σε όλα τα θέματα, νομική βάση κλπ, αφού εσείς μπορεί να τα γνωρίζετε πολύ καλά, αλλά θέλω να υπογραμμίσω ότι ε, αυτή η χρονική στιγμή είναι πολύ σημαντική και το έργο σας είναι πολύ σημαντικό εδώ, ε, να πιέσουμε ούτως ώστε οι νομικές υποχρεώσεις να υλοποιηθούν. Και δεν πρόκειται μόνο για νομικές υποχρεώσεις, αλλά και πολιτικές δεσμεύσεις. Μεταξύ αυτών, πολύ σημαντική είναι η στόχη βιώσιμης ανάπτυξης που ε, έχουν αναλάβει η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι μια ακόμα σημαντική βάση για αυτή τη δουλειά. Για να δούμε τώρα για τι θέμα θα μιλήσω. Δυστυχώς όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια μακρά παράδοση φορολογικών πολιτικών που δεν λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου. Υπάρχουν πολλά θέματα όμως που επηρεάζουν το, η διάσταση του φύλου κοινωνικο-οικονομικά. Και εσείς κυρία Πρόεδρε αναφέρατε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Δηλαδή της, τη διασύνδεση της φορολογίας, κυρίως εισοδήματο και των κινήτρων για να μπουν στην αγορά εργασίας και οι γυναίκες. Δεν θα μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτό το θέμα γιατί ξέρω ότι υπάρχουν αρκετά στοιχεία και έχει αποκτηθεί γνώση επί του θέματος εδώ. Ένα άλλο θέμα είναι οι μειωμένοι συντελεστές για τον ε, φόρο ΦΠΑ ε, και φοροαπαλλαγές σε σημαντικούς τομείς για τις γυναίκες. Εγώ θέλω να διευρύνω την, ε, τις απόψεις μας σχετικά με το θέμα για να συμπεριλάβουμε γενικότερα θέματα και εστιάσεις που πρέπει να μας απασχολήσουν κατεπηγόντως θα παρουσιάσω επτά ζητήματα, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου. Το πρώτο θέμα αφορά το πολύ σημαντικό ευρωπαϊκό εξάμεινο που δομεί τις ευρωπαϊκές πολιτικές μέσα σε ένα χρόνο και προετοιμαζόμενοι για την ομιλία αυτή Έκανα μία ανάλυση των συστάσεων για κάθε χώρα που αφορούν φορολογικά θέματα και αυτό που βλέπουμε είναι ότι όσοι επιτοπλίστων δεν λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου. Ως επιτοπλίστων λέω, γιατί πρόσφατα στην καινούρια πρόταση της Κομισιόν για τις συστάσεις για κάθε χώρα, το θέμα των κινήτρων για την αγορά εργασίας έχει συμπεριληφθεί ή τα αντικίνητρα, αν θέλετε, για τον δεύτερο εργαζόμενο μέσα σε μια οικογένεια. Εκτός αυτού όμως, επί άλλων φορολογικών προτάσεων, δεν λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου. Και οι συστάσεις για κάθε χώρα, ε, ε, εν μέρη τουλάχιστον, συνεπάγονται κινδύνους για την διάσταση του φύλου. Γιατί οι συστάσεις περιλαμβάνουν και προωθούν μετατοπίσεις στη δομή των φόρων που μπορεί να ε, δημιουργήσουν σφάλματα σε ό,τι αφορά τη διάσταση του φύλου και μπορεί να αυξήσουν τις ανισότητες. Τώρα δεν υπάρχει όμως ε, εστίαση στις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι προτάσεις για τα δύο φύλλα. Δεν έχει γίνει μια ανάλυση. Οπότε υπάρχει εδώ μεγάλο πεδίο δράσης. Ένα σημαντικό θέμα και περνώ στο δεύτερο θέμα μου είναι όλη η πορεία που ακολουθεί η φορολογική πολιτική που όλο και περισσότερο στηρίζεται στην έννοια της φορολογίας φιλικής προς την ανάπτυξη. Εδώ θα ήθελα να πω ότι αυτό συνεπάγεται ένα σφάλμα, αν θέλετε, γενέσεις ό,τι αφορά τη διάσταση του φύλου. Γιατί? Γιατί η φορολογία που προσανατολίζεται προς την ανάπτυξη εστιάζει πάρα πολύ στην μείωση του, εταιρι, του εταιρικού φόρου και το είδαμε αυτό στις συστάσεις, περιλαμβάνει και μείωση στο φορολογικό συντελεστή για τις επιχειρήσεις ε, συνολικά και ε, θέλει αύξηση των φόρων κατανάλωσης, ιδιαίτερα του φόρου ΦΠΑ. Δεν είναι καινούριο αυτό. Το έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια ε, μέσα από τις συστάσεις που διατυπώνονταν και που πέρασαν σταδιακά σε αύξηση του, του φόρου του ΦΠΑ και τη χρήση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ και σε φόρους ακίνητης περιουσίας. Δεν θα συζητήσω το αν ε, η φορολογία φιλική προς την ανάπτυξη όντως προωθεί την ανάπτυξη. Γιατί υπάρχουν πολλές προϋποθέσεις εδώ που αφορούν την ελαστικότητα της ζήτησης εργασίας και της προσφοράς εργασίας. Υπάρχουν θέματα μακροοικονομικών προϋποθέσεων και συνθήκων, αλλά τουλάχιστον βάζω ένα ερωτηματικό στο θέμα αυτό της άμεσης συσχέτισης μεταξύ μείωσης εταιρικού φόρου και φόρου εισοδήματος και πέρασμα στο φόρο ΦΠΑ που αυξάνεται. Ιδιαίτερα αν δούμε αυτό το θέμα ε, διαχρονικά Ε, μπορούμε να διατυπώσουμε κάποιες αμφιβολίες για το αν προωθείται η ανάπτυξη. Σίγουρα η φορολογία αυτή δεν αυξάνει ε, την ε, βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του κόσμου, γιατί μεταξύ άλλων δημιουργεί και εισοδηματικά κενά. Δεδομένων των ε, δομών που υπάρχουν και που αφορούν τα δύο φύλλα, αυτή η μετατόπιση στους φόρους ε, επηρεάζει την κατάσταση των δύο φύλων και με βάση τα στοιχεία που έχουμε αυξάνεται έτσι η ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Μία πρόκληση εδώ αφορά την ανάγκη για στατιστικά στοιχεία. Δεν είναι αρκετά. Ούτε έχουμε αρκετά διαθέσιμα στοιχεία σε σχέση με την, ε, τα περιουσιακά στοιχεία και τα εισοδήματα των δύο φύλων. Είναι περιορισμένα τα στατιστικά στοιχεία. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα μπορούσε να πει κανείς, αφού συλλέγει στατιστικά στοιχεία για και περιουσιακά στοιχεία ε, και άλλα εισοδήματα, να συμπεριλάβει τη διάσταση του φύλου και να έχει μια στατιστική βάση για περαιτέρω έρευνα έτσι. Τρίτο σημείο που θέλω να θίξω. Πρέπει να δούμε τα φορολογικά θέματα και την πλευρά των δημοσίων δαπανών ως ένα ενιαίο ζήτημα. Δύο πλευρές του ιδίου νομίσματος. Οι τωρινές τάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπουμε ότι περιορίζουν το δημοσιονομικό χώρο. Άρα υπάρχουν λίγες πηγές διαθέσιμες για τις δημόσιες πολιτικές. Γεννάται το ερώτημα από τη διάσταση των φύλων, μέσα από αυτό το πρίσμα δηλαδή. ποια είναι τα έσοδα που δημιουργούνται συνολικά, ποιος είναι ο δημοσιονομικός χώρος, πόσα έσοδα υπάρχουν για τις απόλυτα αναγκαίες δημόσιες δαπάνες, γιατί και ε, από την πλευρά ενός προοδευτικού φορολογικού συστήματος, αλλά και, και αυτό είναι πιο σημαντικό, από την πλευρά των δημοσίων δαπανών, μπορεί να υπάρξει πολύ μεγάλη συνεισφορά στις ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων. Επίσης, οι προτάσεις μείωσης των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης των εργοδοτών, πρώτον, δεν είναι βέβαιο ότι όντως οδηγούν σε αύξηση της απασχόλησης, γιατί όπως είπα πάντα υπάρχει ένα ερωτηματικό σε σχέση με τις συνθήκες που επικρατούν κάθε φορά στην αγορά εργασίας, αλλά κατά δεύτερο ε, λόγο ε, γίνεται και διάβρωση της φορολογικής βάσης για τα ε, συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Και αυτό πάλι με τη σειρά του οδηγεί σε προβλήματα ανισοτήτων. Ένα άλλο θέμα, να το προσθέσω εν συντομία, γιατί συχνά το ξεχνάμε. Προφανώς είναι πολύ σημαντικό να πάμε προς μια φορολογία φιλική προς το περιβάλλον. Αλλά δεν μπορεί να υποθέσουμε ότι αυτή θα είναι ουδέτερη ως προς τα φύλλα. Αντίθετα, υπάρχει λίγη έρευνα αν και υπάρχει λίγη έρευνα, υπάρχουν κάποιες μελέτες εν που δείχνουν ότι η φορολογία αυτή επηρεάζει τα δύο φύλλα. Άρα είναι ένα θέμα που πρέπει περαιτέρω να εξεταστεί και να συμπεριληφθεί. Ε, προφανώς ε, ε, επηρεάζει το εισόδημα και η διανομή του, αλλά σημαντικά είναι και τα έσοδα και το πώς δομούνται οι πολιτικές μετριασμού και τι σφάλματα ως προς τα φύλλα περιέχουν αυτοί. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη λοιπόν για ανάλυση ε, μέσα από το πρίσμα των δύο φύλων όταν σχεδιάζομαι οικολογική φορολογία. Αλλαγή της φορολογικής δομής, αυτό είναι το πέμπτο σημείο, και προτάσεις για μεταρρύθμιση που θα προωθήσει ένα πιο δίκαιο φορολογικό σύστημα, πιο ισότιμο. Τα πιο προοδευτικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένης της εταιρική και φορολογίας και της φορολογίας προσωπικού εισοδήματος, δημιουργούν ανισότητες ε, όπως και ο φόρος ε, κληρονομίας και οικονομικών, δημοσιο... Ε, χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Γνωρίζουμε ότι χρειάζεται να σταματήσουμε την φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή, αλλά και αυτή η προσπάθεια ενέχει μια διάσταση του φύλου, διότι και εδώ υπάρχει μεγάλη ανισότητα σε ό,τι αφορά την κατανομή του πλούτου και τις δομές της ιδιοκτησίας. Προχωρώ στις δύο τελευταίες μου θέσεις που είναι πιο πολιτικές αν θέλετε. Πρώτον, βάσει της παρατήρησης ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την φορολογική πλευρά του αλλά και γενικότερα, ε, δεν ενσωματώνει παρά μόνο λίγο την διάσταση του φύλου και η Κομισιόν το ξέρω έχει αρχίσει να δουλεύει πάνω σε αυτά τα θέματα. Αυτό που προτείνεται είναι μια τακτική ε, ανάλυση αξιολόγηση αντικτύπου ε, στα δύο φύλλα ε, και πάνω σε αυτή τη βάση να γίνουν αλλαγές και να υπάρχουν τα στοιχεία αυτά ως βάση για βελτιωτικές προτάσεις στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Όμως δεν πρόκειται μόνο για την αξιολόγηση του αντίκτυπου στα φύλλα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί και γνώση των οικονομικών που αφορούν τα δύο φύλλα σε όλη τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν μερικές ομάδες που υπάρχουν ε, ορισμένα ε, στοιχεία που πρέπει να ενσωματω που υπάρχουν στη διάθεσή μας και θα πρέπει να τα συμπεριλάβουμε. Οι στόχοι που αφορούν το φύλλο θα πρέπει να ενσωματωθούν σε όλα τα ε, κείμενα της διαδικασίας, αρχίζοντας από την ετήσια ε, έκθεση για την ανάπτυξη μέχρι τις ε, συστάσεις για κάθε χώρα χωριστά. Και αυτό σημαίνει ότι και το Κοινοβούλιο θα έχει μεγαλύτερο λόγο σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ιδιαίτερα θα ε, αναβαθμιστεί ο ρόλος της δικής σας ε, σεβαστής επιτροπής ε, για να εντάξει τη διάσταση του φύλου. Τέλος θα κάνω μια πρόταση η οποία είναι κάπως πιο μακροπρόθεσμη και αφορά τις θεσμικές καινοτομίες. Επειδή μέχρι τώρα αγνοεί το θέμα της ισότητας των φύλων, ιδιαίτερα στις οικονομικές πολιτικές και ακόμα περισσότερο στα φορολογικά θέματα, προτείνω να δημιουργηθεί ένα συμβούλιο α, ισότητας των φύλων και φορολογικής πολιτικής, το οποίο θα λειτουργεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο κρατών μελών ως πηγή γνώσης, δημιουργίας ικανοτήτων και πηγή παροχής ανεξάρτητης ε, εμπειρογνωμοσύνης και συμβουλών. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίασή σας και τώρα θέλω να δώσω το λόγο στον κύριο Βαντάμ που είναι από το Βέλγιο, πρόεδρος ε, του Friday Group. Είναι σύμβουλος για θέματα υγείας και κοινωνικά ε, στον Πρωθυπουργό του Βελγίου και είναι μέλος του Συμβουλίου, του Διεθνού Συμβουλίου μάλλον, για θέματα υγείας και κοινωνικά θέματα. Παρακαλώ. Good Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, για την ευκαιρία αυτή που μου δίνετε. Ήμουν αναπληρωτής επικεφαλής του προσωπικού του Πρωθυπουργού το καλοκαίρι που μας πέρασε. Αλλά η γυναίκα μου που είναι από την Νορβηγία ε, βρήκε δουλειά στην Νορβηγία και τελικά πήγαμε εκεί. Και τον τελευταίο χρόνο είμαι εκεί στην Νορβηγία. Βέβαια πάντα δουλεύω ως πρόεδρος στο Friday Group και υπό αυτή την ιδιότητα βρίσκομαι σήμερα μαζί σας. Ποιοι είμαστε λοιπόν. Είμαστε ένα πλουραλιστικό think tank για νέους. Είμαστε και μέρος του Ιδρύματος ε, του Βασιλιά Μπούντουε και τον Δεκέμβριο είχαμε μία έκθεση την οποία και θα σας παρουσιάσω για 10-15 λεπτά σήμερα που έγραψα από κοινού με την Μαρίκα Άντερσον και την Αταλή Φρανσουά, που δεν μπορούν να είναι μαζί μας σήμερα. Λοιπόν, περί τίνος πρόκειται. Αρχίζουμε με μία παρατήρηση. Και αυτή είναι ότι ακόμα και εμείς, που είμαστε πολύ γενναιόδοροι σε αυτό, δεν καταφέραμε να έχουμε τόσες γυναίκες όσες θα θέλαμε όσους και άντρες. Και γιατί είναι τόσο δύσκολο να βρει κανείς γυναίκες και γιατί οι γυναίκες υποαντιπροσωπεύονται στο δημόσιο βίο. Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι το θέμα της ανισότητας απέναντι στο χρόνο είναι το ζήτημα. Σήμερα διαπιστώνουμε ότι οι γυναίκες κάνουν πολύ περισσότερη απλήρωτη δουλειά από όσο κάνουν οι άντρες. Στο Βέλγιο κάθε μέρα κατά μέσο όρο οι γυναίκες μια μισή ώρα παραπάνω δουλεύουν με απλήρωτη εργασία από ότι οι άντρες, που σημαίνει τρεις μήνες το χρόνο απλήρωτη εργασία. Άρα λοιπόν χάνουν και πολλά εισοδήματα. Και εξού και δεν αντιπροσωπεύονται παρκώς στο δημόσιο βίο. Και υπάρχει τέτοια διαφορά στους μισθούς και στις συντάξει. Οι γυναίκες λοιπόν χρησιμοποιούν το χρόνο τους διαφορετικά από ό,τι άντρες. Και αυτό με το που έρχονται και τα παιδιά γίνεται ακόμα χειρότερο. Και σε αυτό θα επικεντρωθώ σήμερα. Πώς δηλαδή μπορούμε, πώς θα μπορούσαμε να προσφέρουμε περισσότερη ισότητα απέναντι στο χρόνο στα δύο φύλλα. Θα επικεντρωθώ λοιπόν στο Βέλγιο, μια που είναι μια περίπτωση που γνωρίζω καλά και που κάναμε διάφορες μεταρρυθμίσεις για να αντιμετωπίσουμε τα κοινωνικά επιδόματα και τις φορολογικές πολιτικές ανάλογα. Αυτή είναι η εικόνα. Τώρα, Υπάρχουν και μερικά καλά νέα, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως γνωρίζετε, ξεκίνησε τον Απρίλιο με την αναθεώρηση της ε, οδηγίας για την ε, γονική άδεια. Γιατί είναι λοιπόν σημαντικό να επενδύουμε στις φορολογικές πολιτικές και σε άλλα μέτρα. Αυτό θα εξηγήσω τώρα και θα καταλήξω και σε μια συγκεκριμένη πρόταση για το Βέλγιο. Τώρα όσον αφορά την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο θέμα αυτό της ανισότητας μεταξύ των δύο φύλων. Προσφέρει μια γενικότερη και καλύτερη γονική άδεια. προτείνει τέσσερις μήνες γονική άδεια για τα ζευγάρια που θα πληρώνεται σε επίπεδο αναρωτικής άδεια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και φυσικά προβλέπεται ευελιξία Και γιατί είναι καλό αυτό. Και γιατί δεν λύνει και το πρόβλημα πλήρως. Η χώρα μου λοιπόν, το Βέλγιο, θεωρείται προδευτική σε αυτά τα ζητήματα. Θεωρεί τον εαυτό της κάπως προδευτικό. Είναι κάπου στη μέση βέβαια μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Αν λοιπόν εγκρίνονταν και από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο η οδηγία αυτή, τότε η εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα προχωρούσε, θα κέρδιζε έδαφος και θα πήγαινε πιο κοντά στις πιο προδευτικές χώρες. Δεύτερον, δεν γίνεται τίποτα όσον αφορά το φορολογικό. Και είναι και αυτό ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Οπότε, ναι, δεν έχει λυθεί το πρόβλημα και γι' αυτό συνεχίζουμε τώρα. Γιατί είναι τόσο σημαντική η γονική άδεια διαμητρότητα πατρότητα. Γιατί έτσι αυτή η απλήρωτη εργασία κατανέμεται περισσότερο δίκαια, περισσότερο ισότιμα υπάρχουν ε, πατέρες οι οποίοι από την αρχή με το που γεννιούνται τα παιδιά τους, ασχολούνται με τα παιδιά τους, αναλαμβάνουν αυτή την απλήρωτη εργασία, κάνουν πολλές δουλειές στο σπίτι μέχρι το τέλος της ζωής τους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να υπάρχει αυτή η ισορροπία, δηλαδή αυτή η απλήρωτη εργασία να κατανέμεται ισότιμα ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες. Με αυτόν τον τρόπο οι άντρες εμπλέκονται περισσότερο στον ιδιωτικό βίο, πράγμα το οποίο συγχρόνως επιτρέπει στις γυναίκες να επενδύουν περισσότερο στο δημόσιο βίο και άρα να μειώνεται και η διαφορά στους μισθούς. Οι έρευνες εξάλλου έχουν δείξει ότι τα παιδιά τα οποία ε, μεγαλώνουν με τους πατεράδες τους στην αρχή στο σπίτι και γενικά που οι πατεράδες αναλαμβάνουν όλο και περισσότερη δουλειά στο σπίτι, μεγαλώνουν καλύτερα και έχουν ε, καλύτερα, καλύτερη εικόνα για την ισορροπία στο σπίτι. Και το έχουν πει και σε πολλές υπηρεσίες πατεράδες που ό,τι θέλουν να συμμετέχουν περισσότερο ε, στη δουλειά στο σπίτι και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα από τις έρευνες πάντα αποδεικνύεται αυτό ότι οδηγεί σε λιγότερα διαζύγια. Και βέβαια και σε μεγαλύτερη παραγωγικότητα, γιατί έτσι οι γυναίκες συμμετέχουν περισσότερο στην αγορά εργασίας. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό αυτό. Όμως, πώς θα πιέσουμε για περισσότερη ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Είπαμε, η γονική άδεια είναι κάτι πολύ σημαντικό ήδη. Όμως, όπως έχει πει ήδη από το 12 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν έρθει η στιγμή άντρες και γυναίκες να πάρουν την απόφαση να φτιάξουν μια οικογένεια, δεν αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο τις επιλογές τους. Δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες όπως είπε και συνάδελφος. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που πρέπει να κοιτάξουμε, σας είπα το ένα είναι η γονική άδεια, το άλλο είναι η φορολογία. Το πρώτο. Πώς λοιπόν μπορούμε να έχουμε φιλικές προς την οικογένεια πολιτικές χωρίζουμε τις χώρες σε τέσσερις κατηγορίες και τελικά μόνο οι σκανδιναβικές χώρες, οι βόρειες χώρες έχουν πραγματικά πολιτικές υπέρ της οικογένειας που να αντιμετωπίζουμε τον ίδιο τρόπο τους άντρες και τις γυναίκες. Για τις άλλες χώρες μέλη υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Φορολογικές τώρα επιλογές. Η κυρία Γκούνεσον που θα μιλήσει μετά από μένα έχει αναλύσει το θέμα ήδη από το 2016 και λέει ότι μόνο η Σουηδία και η Φιλανδία έχουν καταφέρει να έχουν ένα καλό φορολογικό σύστημα. Πράγμα που σημαίνει ότι σε όλες τις άλλες χώρες υπάρχουν διατάξεις που τελικά δίνουν κίνητρα σε έναν από τους δύο γονείς να επωφεληθεί από την φορολογία και όχι και τους δύο. Κάτι το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές οι γυναίκες που κερδίζουν λιγότερα συνήθως σήμερα να είναι αυτές οι οποίες ε, τελικά δεν επωφελούνται από φορολογικές ελαφρύνσεις. Άρα ότι και αυτό είναι υπέρ της ισότητας. Πρέπει λοιπόν να γίνει αναθεώρηση της γονικής άδειας από τη μια είπα φορολογία, από την άλλη κάτι που γίνεται σε επίπεδο χωρών μελών. Οπότε το ζήτημα είναι πώς θα προσπαθήσουμε να τα υλοποιήσουμε αυτά πολύ συγκεκριμένα. Αν κοιτάξετε το πρώτο θέμα, την γονική άδεια και την άδεια και πάλι αν κοιτάξουμε τι γίνεται στο Βέλγιο, διαπιστώνουμε ότι είναι οι γυναίκες εκείνες οι οποίες πιο συχνά χρησιμοποιούν τη δυνατότητα αυτή για γονική άδεια τα δύο τρίτα της γονικής άδεια ε, πηγαίνουν σε γυναίκες, γιατί οι γυναίκες τις ζητάνε. Αν λοιπόν θέλουμε περισσότερη ισότητα απέναντι στον χρόνο, πρέπει να δώσουμε κίνητρα στους άντρες να χρησιμοποιούν και αυτοί εξίσου τη δυνατότητα αυτή στη γονική άδεια. Και αυτό κάναμε και στο Βέλιο. Και γι' αυτό και αρχίσαμε με την οδηγία αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τα μπρος, αλλά εξακολουθεί να έχει κάποια προβληματάκια. Έτσι λοιπόν προχωρούμε σε μία πολύ συγκεκριμένη μεταρρύθμιση για το σύστημα της γονικής άδειας και άδειας πατρότητας στο Βέλιο. Τέσσερις μήνες γονική άδεια επιτρέπουμε που πληρώνεται με 700 ευρώ το μήνα. Βέβαια δεν φτάνουν τα χρήματα αυτά ώστε να αποτελούν κίνητρο ώστε οι άνθρωποι, κυρίω οι άντρε να ζητήσουν τη γονική άδεια. Από την άλλη μεριά, βέβαια, δικαιούνται οι πατεράδε 10 μέρε κάτι το οποίο θα ήταν καλό να ισχύει παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, επειδή είμαι και εγώ από την πολιτική, Καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι αυτά τα ζητήματα και περίπλοκα. Γι' αυτό και προσπαθούμε να σχεδιάσουμε μια μεταρρύθμιση της γονικής άδεια που να δίνει κίνητρα στους άντρες να παίρνουν τη γονική τους άδεια όσο γίνεται πιο γρήγορα. Δηλαδή αμέσως μετά τη γέννηση του παιδιού, αν αρχίσει ο άντρας να ασχολείται με το παιδί του, τότε διαπιστώνουμε ότι και στη συνέχεια θα αναλαμβάνει όλο και περισσότερα καθήκοντα στο σπίτι. Οπότε πρέπει από τη μια μεριά ε, να αποφέρει η γονική άδεια αρκετά χρήματα και στους πατεράδες και από την άλλη μεριά να τους είναι και ελκυστική. Τέσσερις μήνες λοιπόν μπορούν να πληρώνονται οι άντρες με 700 ευρώ το μήνα. Αυτό λέμε υπάρχει ήδη. Αλλά αν αυτούς τους τέσσερις μήνες λέμε τους πάρεις αμέσως μετά την γέννηση του παιδιού σου, τότε έχεις δικαίωμα όχι μόνο αυτά στους τέσσερις μήνες επί 700 ευρώ, αλλά πέντε φορές 700 ευρώ μέσα σε τρεις μήνες. Δηλαδή λίγο πολύ δια, διπλασιάζουμε τις απολαβές για δυόμιση μήνες. Οι πατεράδες, τα νοικοκυριά μπορούν να αυξήσουν κατά 700 ευρώ τα έσοδά τους, κάτι το οποίο μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για να ασχοληθούν με τα παιδιά οι πατεράδες. Δέκα μέρες λοιπόν άδεια μετά τη γέννηση και στη συνέχεια γονική άδεια, την αναθεωρημένη, δυόμισι μήνες δηλαδή με 1500 ευρώ το μήνα. Άρα πρόκειται τελικά για τρεις μήνες κατά τους οποίους μπορεί να μείνει σπίτι ο πατέρας να ασχοληθεί το παιδί του με μια αρκετά αξιοπρεπή αμοιβή. 1500 ευρώ το μήνα δηλαδή, κάτι το οποίο θα ήταν αρκετό πιστεύουμε για να αποτελέσει κίνητρο για τους πατεράδες να μείνουν στο σπίτι και να χρησιμοποιήσουν αυτή τη γονική άδεια, τη μεταρρυθμισμένη. είναι λίγο πολύ όπως στις σκανδιναβικές χώρες. Ποιο είναι το κόστος αν λάβουμε υπόψη μας και φορολογικές και μη φορολογικές. Πρόκειται για 15.000 ευρώ. Με 11 εκατομμύρια κατοίκους 15 εκατομμύρια στοιχίζει τελικά. Τώρα πώς θα το χρηματοδοτήσουμε αυτό. Όπως και σε άλλες χώρες έχουμε φορολογικά μέτρα τα οποία διευκολύνουν ε, τους ε, συζύγους, τους συντρόφους, αν ένας από τους δύο μείνει στο σπίτι, έχει κάποιες φορολογικές ελαφρύνσεις. 10.200 ευρώ το χρόνο. Είναι ένα κίνητρο, κυρίως για τις γυναίκες όμως προς το παρόν, να μείνουν σπίτι. Πολλές αρχές, το ακούσαμε, είναι κατά αυτών των φορολογικών μέτρων. βασικά βασιζόμαστε σε αυτό που ονομάζουμε marital quotient. 600 εκατομμύρια το χρόνο που χρησιμοποιούνται για να χρηματοδοτείται η γονική άδεια και η άδεια πατρότητας. Γνωρίζω βέβαια ότι δεν είναι πάντα εύκολο για τους πολιτικούς και τα περισσότερα συντηρητικά κόμματα εδώ στο Βέλγιο, αν με τι άλλο, Τι θέλουν αυτή την φορολογική απαλλαγή. Αν καταργηθεί θα ήταν δύσκολο και μη ρεαλιστικό ίσως, οπότε εμεί λέμε να μην υπάρχει αναπροσαρμογή όπως μπορείς να κάνεις στο τέλος της χρονιάς κάθε φορά. Αλλά πιο αρεά. Αυτό είναι κάτι αρκετά ρεαλιστικό πιστεύω. Και που θα οδηγήσει αυτό θα βοηθήσει και τις γυναίκες και τους άντρες να προσφεύγουν πιο συχνά οι ίδιοι στη γονική άδεια. Προχωρούμε επίσης σε προτάσεις για χαμηλότερο ΦΠΑ σε διάφορα προϊόντα, υγιεινής και άλλα. Ποιες είναι οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Είναι μερικά πράγματα τα οποία συχνά τα ξεχνάμε. Πρώτα απ' όλα, τι γίνεται με τους ελεύθερους επαγγελματίες, που συχνά τους ξεχνάμε. Τι γίνεται με τις περιπτώσεις αναδοχής, με τις ανάδοχες οικογένειες, ανάδοχους γονείς, οι οποίοι δεν δικαιούνται όπως και οι βιολογικοί γονείς, τη γονική άδεια, άδεια μητρότητας, πατρότητας κλπ. Αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί για την άδικο. Και τρίτον, η οδηγία της Επιτροπής που θα υποβληθεί στο Κοινοβούλιο σύντομα, από ό,τι καταλαβαίνω, προβλέπει στο άρθρο 8 ότι τέσσερις μήνες γονικής άδειας δεν μπορούν να μεταφερθούν στον άλλον ε, εταίρο ή να αποζημιωθούν σε επίπεδα αναρωτικής άδειας. Το οποίο είναι πολύ χειρότερο από αυτό που ισχύει στο Βέλγιο σήμερα. Και φοβάμαι ότι αυτό θα είναι το βασικό που θα συζητηθεί και στο Συμβούλιο. Και μπορεί τελικά το άρθρο αυτό να μην περάσει. Οπότε θα έλεγα και εσείς να πιέσετε ώστε το άρθρο 8 να παραμείνει. Και για την άδεια μητρότητας, για την οδηγία αυτή, θα έπρεπε επίσης να αναθεωρηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να γίνει πιο γενναιόδορη. για να γίνονται οικογενειακοί δεσμοί ακόμα πιο στενοί. Βασιζόμαστε σε εσά λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Τώρα περνάμε στην επόμενη μελέτη. Θα δώσω το λόγο. Εσσα Γκούναρσον από τη Σουηδία. Η κυρία Εσσα Γκούναρσον έχει συνεισφέρει και σε εθνικό επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο ασχοληθεί με την εκπαίδευση και τις νομικές ρυθμίσεις και το ρόλο που παίζουν στην ισότητα των φύλων. Σας ευχαριστώ, λέει η κυρία Γκούναρσον, για την δυνατότητα που μου δώσατε να πάρω μέρος στη συγγραφή αυτής της έκθεσης. Είναι, θα έλεγα, μία πρόκληση του να εφαρμόσει κανείς την προοπτική του φύλου στο θέμα της φορολογίας, ιδιαίτερα στον τομέα των νομικών ρυθμίσεων και των κανονισμών για την φορολογία. Είναι ένα θέμα πραγματικά ε, mainstream, το οποίο για πάρα πολλούς πολιτικούς και πάρα πολλούς πολίτες ε, παρουσιάζει τεχνικά χαρακτηριστικά και είναι ένας τομέας μερικές φορές όπου η κατανόηση και η γνώση δεν είναι σαφής. Αυτό το οποίο προσπαθώ λοιπόν να κάνω είναι να δώσω κάποιες εξηγήσει και για τη φύση της φορολογίας σαν δραστηριότητα και να εφαρμόσουμε φυσικά κάνοντας το αυτό <clears throat> την προοπτική του φύλου. Βλέπετε εδώ τους ε, συγγραφείς της έκθεσης και οι τρεις Είμαστε ερευνητές στο πρόγραμμα του Horizon 2020, του οποίου είμαι συντονίστρια, το Fairtax. Είναι ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια και θα τελειώσει στο τέλος, στις αρχές μάλλον του 19 στα πλαίσια της προβληματικής κοινωνικών προκλήσεων. Αυτά για τα τυπικά. Πρόκειται για μια έρευνα την οποία υποστηρίζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία συμμετέχει σε ένα τμήμα της ομάδας για το Fairtax Βλέπετε ότι είναι και η Ούλρικε Σπάγκεμπερκ. Είναι φεμινίστριες πανεπιστημιακές, όχι μόνο σε θέματα φεμινιστικών σπουδών, αλλά ασχολούνται πολύ ε, με θέματα φορολογίας και με θέματα ε, προβληματικής γύρω από το φύλλο. Αυτή είναι η στόχη του προγράμματος. Να πω ότι κάνουν αρκετά πράγματα τα οποία δεν ε, εξετάζονται από πλευράς ε, ε, προοπτικής φύλου, αλλά σε επίπεδο γνωστικό προσπαθούμε να εντάξουμε την προβληματική του φύλου όποτε αυτό είναι εφικτό και όποτε είναι φυσικά σχετικό. Αυτό είναι ένα αίτημα θα έλεγα το οποίο έχουμε και προς τα ευρωπαϊκά όργανα η προβληματική του φύλου στον τομέα της φορολογικής δραστηριότητας δεν θα πρέπει να θεωρηθεί σαν κάτι το εξωτερικό, σαν κάτι το δευτερεύον, όταν γίνονται συζητήσεις για την φορολογία στα κράτη-μέλη <clears throat> και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην έκθεση λοιπόν μπορείτε να δείτε κάποια βασικά ευρήματα θεωρούμε ότι η ισότητα των φύλων είναι κομβικό θέμα σχετικά με την βιωσιμότητα των πολιτικών των ευρωπαϊκών στο μέλλον. Και αυτό ισχύει για όλες τις συζητήσεις οι οποίες γίνονται στον τομέα της φορολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. λέμε στην έκθεση ότι οι πολιτικές αυτές οι φορολογικές έχουν μία θα έλεγα αναδιαναμετική ε, προοπτική όπως επίσης και μία προσπάθεια κατανομής των ευθυνών ε, ανά τομέα. Ένα απλό μήνυμα εδώ είναι ότι το φορολογικό σύστημα δείχνει σε μια πρώτη φάση <clears throat> τις γυναίκες φτωχότερες από ό,τι είναι μερικές φορές και συνεπώς έτσι δεν βοηθά τις γυναίκες να αναπτύξουν την οικονομική τους ανεξαρτησία. Λειτουργεί διαβρωτικά ως προς την οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών. Ε, βιώσαμε μία μακρά περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας η κοινωνικο-οικονομική πραγματικότητα λειτουργεί ως υποκείμενο της κυριαρχής κατάστασης για τις γυναίκες. Το φορολογικό σύστημα, με λίγα λόγια, δεν έχει βοηθήσει να βγουν οι γυναίκες από τις παγίδες της ένδυας. Δεν έχει βοηθήσει το φορολογικό σύστημα να μειωθεί η διαφορά στα εισοδήματα. Δεν έχει βοηθεί να καλυφθούν οι ανισότητες στον τομέα της πρόνοιας και δεν έχει βοηθήσει να κλείσει κάπως, να μειωθεί το επίπεδο πλούτου ανδρικού από τη μία και γυναικείου από την άλλη. Η προβληματική του φίλου λοιπόν γενικά είναι απαραίτητη. Όπως ακούσαμε από την Ελισάβετ, έχουν υπάρξει πολλές μελέτες τις οποίες ελέγχουν ε, τα ευρωπαϊκά όργανα για τη σχέση ανάμεσα στην φορολογία, τα φορολογικά συστήματα δηλαδή, και τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούν αντικίνητρα για τον ρόλο των γυναικών στην αγορά εργασίας. Η Ελίζαμπεθ έχει υπογραμμίσει επίσης ότι τα όργανα της Ένωσης και τα κράτη-μέλη δεν σέβονται τις νομικές υποχρεώσεις τις οποίες έχουν αναλάβει και δεν έχουν μπορέσει να διασφαλίσουν μια ουσιαστική φορολογική ισότητα. Αυτά τα έχει παρουσιάσει γραπτά η Ελισάβετ. Θα ήθελα όμως εδώ να υπογραμμίσω την λέξη διασφαλίζω, η οποία θα πρέπει να είναι ο βασικός ρόλος των ευρωπαϊκών οργάνων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως και των διοικήσεων των κρατών μελών. Μπορεί βέβαια κάποιος να πει ότι δεν είναι ένας από τους κατεξοχήν πολιτικούς τομείς παρέμβασης της Ένωσης, μιας και είναι εθνική πολιτική αλλά όταν είμαστε υποχρεωμένοι να διασφαλίσουμε ακριβώς ε, την παρουσία και την ισχύ των αρχών αυτών σε όλους τους τομείς και δεν θα πρέπει να μην ισχύει αυτό για την φορολογία. Συνεπώς λοιπόν υπάρχουν ανηλυμένες υποχρεώσεις επί των οποίων μπορούμε να εργαστούμε και νομίζω ότι και εσείς στην Επιτροπή σας τις γνωρίζετε αυτές τις υποχρεώσεις, αλλά σαν καθηγήτρια δικαίου θέλω να επιμείνω σε αυτήν την θεμελιώδη θα έλεγα παρατήρηση την οποία έκανα, έτσι ώστε να μπορέσουμε χρησιμοποιώντας τη βασική αυτή αρχή να σημειώσουμε προόδο προς την ισότητα σε επίπεδο φόρων. Εδώ βλέπετε κάποια ποσοτικά στοιχεία τώρα για τη δομή της φορολογίας που υπογραμμίζουμε στην έκθεση που έχουμε παρουσιάσει. Δείχνουμε το πού βρισκόμαστε στην παρούσα φάση σχετικά με τα φορολογικά έσοδα γενικότερα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπετε ότι εξαρτώμεθα εμπολής από το εισόδημα των μισθωτών κυρίως, από τους μισθούς δηλαδή, όπως επίσης και από εργαζομένους γενικότερα σε μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις για τις γυναίκες. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε πρόβλημα σε σχέση με τη φορολογία του κεφαλαίου όπως επίσης και στον τομέα των φορολογικών, των περιβαλλοντικών φορολογικών συστημάτων, αλλά κυρίως εξαρτώμεθα από την φορολογία της εργασίας. What I mentioned earlier is that we, during many uh, decades now, have had a, a, a... Κατά τη διάρκεια πολλών δεκαετιών υπήρξε μια ιδεολογία θα έλεγα φορολογική η οποία λειτουργούσε κυρίως αναπτυξιακά. Είχε βοηθήσει να υπάρξει μια ισχυρή βάση στον τομέα των οικονομικών μελετών. Αλλά μετά από τον Πικετή το 2014 οι οικονομολόγοι μετακινήθηκαν λίγο και συνειδητοποίησαν από τον Πικετή και μετά ότι η φορολογία για την ανάπτυξη φαίνεται ότι απονομιμοποιείται αφεαυτής. Δηλαδή ε, γενικά στην κοινωνία υπάρχει ισχυρό ε, φορολογικό φάρος το οποίο λειτουργεί αντιπαραγωγικά σε σχέση με την ανάπτυξη. And as Και όπως είπα νωρίτερα, όταν το αναδιανεμητικό προφίλ αν θέλετε ε, χάνεται μέσα στο εθνικό φορολογικό σύστημα, γίνεται δευτερεύον ε, και επικρατεί η συγκεκριμένη ιδεολογική χρήση της φορολογίας, τίθεται ένα θέμα εδώ, αν πράγματι δηλαδή μπορούμε να στηρίξουμε πλέον τα κράτη πρόνοιας, το κράτος πρόνοιας, αν υπάρχει πλέον μέλλον για το κράτος πρόνοιας γιατί ένα κράτος που έχει ε, τέτοιου είδους πρόνοια πρέπει να έχει και τα αντίστοιχα έσοδα, τους πόρους για να το στηρίξει. Αυτό το οποίο είναι επίσης προφανές ότι έχει υπάρξει μια μετακίνηση του φορολογικού βάρους από τους άνδρες στις γυναίκες. Τι εννοώ. Η φορολογία σε επίπεδο κεφαλαίων σε περιπτώσεις συγκεκριμένες στην Ένωση είναι πάρα πολύ χαμηλή. Στην Σουηδία ας πούμε για κάποια επίπεδα πλούτου έχουμε ένα 20% ενώ σε άλλου τύπου δραστηριότητες έχουμε φορολογικές βάσεις οι οποίες ξεκινούν, φορολογικά ποσοστά που ξεκινούν από το 50%. Εδώ οι γυναίκες όμως φύγονται διπλά, ιδιαίτερα μέσω των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Το χαμηλό επίπεδο επιβολής στο κεφάλαιο είναι κάτι το οποίο ευνοεί τους άνδρες. Αυτή είναι μια απλή κοινωνικο κοινωνικο-οικονομική πραγματικότητα. Και όταν εξετάζουμε το θέμα της ε, φορολογίας εισοδήματος βλέπουμε ότι η, τα ποσοστά της φορολογίας ε, έχουν ε, κατέβει αρκετά. Έχουμε να κάνουμε με ένα σύστημα το οποίο αλλάζει σταδιακά αλλά με πολύ αργή ταχύτητα και σε ορισμένες χώρες μέλη υπάρχει θα έλεγα ένα φορολογικό προφίλ εισοδήματο το οποίο είναι κατά αποκοπήν σταθερό. Τώρα, λοιπόν, τι είναι εύκολο να δει κανείς εδώ. Στην συγκεκριμένη διαφάνεια βλέπει ε, το θέμα των φορολογικών δαπανών και είναι δύσκολο να συλλάβει κανείς. Ε, οι δαπάνες, ε, οι απαλλαγές, οι εκπτώσεις είναι αναπόσπαστα τμήματα του φορολογικού συστήματος. Συνεπώς μπορεί να υπάρχουν επιστροφές σαν παράδειγμα για ιδιωτικές ασφαλείες, συνταξιοδοτικές. Μπορεί να υπάρχουν επίσης ε, φορολογικές ελαφρύνσεις για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις Μπορεί να υπάρχουν επίσης και άλλου τύπου ε, θα έλεγα μειώσεις ε, ε, φορολογικού τύπου οι οποίες δεν είναι όρατες αλλά βάζουν ανώτατα όρια στα έσοδα του κράτους και κυρίως ωφελούν τους άνδρες. Γιατί οι άνδρες είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τα υψηλά εισοδήματα που ωφελούνται και δεν βλέπουμε σαν παράδειγμα την μη αμοιβόμενη εργασία η οποία παρέχεται από τις γυναίκες κυρίως, το συζητήσαμε το θέμα αυτό και στα πλαίσια της γονικής άδειας και αυτό το οποίο έχει σημασία να δει κανείς εδώ είναι ότι αυτά τα αποδιδόμενα εισοδήματα σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό είναι μεν κομμάτια των, ε, των εισοδημάτων από την επιχειρηματικότητα, αλλά κυρίως οι άνδρες είναι αυτοί και πολλές φορές τα τεκμήρια χρησιμοποιούνται κυρίως εις βάρος των γυναικών. Και υπάρχουν πολλές ανισότητες σε επίπεδο νοοτροπίας που είναι βαθιά αγκυρωμένες στα φορολογικά συστήματα. Τώρα για μεμονωμένα, το πρόβλημα μάλλον αν θέλετε ατομικής, έλλειψης ατομικής φορολόγησης. Σε 19 από 28 χώρες μέλη υπάρχει ένα καταποκοπήν ποσοστό. Βλέποντας πιο προσεκτικά υπάρχουν μειώσεις και διευκολύνσεις φορολογικές, επιστροφές και όταν γίνεται μια ατομική αξιολόγηση του φορολογικού συστήματος ελέγχονται ακριβώς τα τεκμήρια τα οποία επηρεάζουν την, τις κοινωνικές παροχές τις οποίες την χάνει το νοικοκυριό, τις οποίες δέχεται το νοικοκυριό. Και υπάρχουν αρκετά συστήματα φορολογικά που λειτουργούν με γνήσιο τρόπο στην Ευρώπη. Εγώ όπως σας είπα έχω ασχοληθεί και με συστήματα φορολογικά και με συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και από την εμπειρία την οποία έχω μέχρι τώρα δεν θα πετύχουμε ισότητα των φύλων στον τομέα αυτό, αν συνεχιστούν τα πράγματα όπως έχουν σήμερα. Έχω ξοδέψει αρκετή ώρα. και θα ήθελα να αναφερθώ τώρα στο, στη φορολογία υψηλών εισοδημάτων Εκεί όπου υπάρχει πρόβλημα στα υψηλά εισοδήματα, αυτό ισχύει και για τη διαφορά των φύλων. Όταν μιλάει κανείς για υψηλά εισοδήματα στη Σουηδία, μιλάει κυρίως για έγκυο ιδιοκτησία. Έχουμε με ένα πολύ μεγάλο κενό, μια πολύ μεγάλη διαφορά και οι μελέτες δείχνουν ότι οι γυναίκες ελέγχουν το, 50, το 15% των ιδιοκτησιών και το υπόλοιπο το ελέγχουν οι άνδρες. Συνεπώς λοιπόν ο πλούτος σορεύεται στους άνδρες και σε σχέση τώρα με τους φόρους κατανάλωσης ε, υπάρχουν και εδώ κάποιες μικρές διαφορές όπως μειώσεις φορολογικών ποσοστών Δεν έχουμε και πάρα πολλά στατιστικά δεδομένα τα οποία να μπορούν να γίνουν αντικείμενο εξέτασης μεμονωμένα με ξεχωριστό τρόπο <clears throat> γιατί χρησιμοποιούμε κυρίως το υπόδειγμα των εισοδημάτων των οικοκυριών. Πάντως, αυτοί οι οποίοι έχουν το υψηλότερο εισόδημα είναι αυτοί που έχουν και τα υψηλότερα επίπεδα πλούτου και σωρεύουν ακόμα περισσότερο αντίστοιχα. Πρέπει λοιπόν να δει ότι η κατανομή των φόρων κατανάλωσης, των φόρων αυτών, θα πρέπει να αναφέρεται στο σύνολο της φορολογικής δραστηριότητας και όχι αυτόνομα και θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο της αλυσίδας της φορολογικής. Είδαμε στην μεταρρύθμιση της φορολογίας το 1991 στη Σουηδία ότι όταν κατέβηκε το, φορο, το ποσοστό επιβολής όταν οι εξαιρέσεις έγιναν περισσότερες και πιο τολμηρές, αυτό λειτουργεί ε, θα έλεγα με τρόπο περιοριστικό για τον υπολογισμό των υπόλοιπων εισοδημάτων. Εμείς περιμένουμε να κάνουμε μια νέα μεταρρύθμιση, η προηγούμενη είναι του 71 σε σχέση με τη φορολογία εισοδήματος. γιατί αλλιώς ο ρόλος των γυναικών είναι ένας ρόλος ο οποίος λειτουργεί ε, πολύ περιοριστικά. Στο τέλος της έκθεσης βλέπετε τις συστάσεις μας. Οι περισσότερες δείχνουν ότι απαιτείται περισσότερη έρευνα, πιο αναλυτικά δεδομένα, και θα πρέπει να υπάρξει ένα σύστημα το οποίο να αναλύει με σωστό τρόπο τις ανισότητες οι οποίες σοβούν στο εσωτερικό του, διαρθρωτικά. Ελπίζουμε ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα αναλάβουν τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουν σύμφωνα με τη συνθήκη και θα αντιμετωπίσουν την πρόκληση προώθησης ακριβώς των σχέσεων ανάμεσα στη φορολογία και την προβληματική των φύλων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την καθηγήτρια Γκούναρσον που μας παρουσίασε τη μελέτη αυτή. Τώρα, περνάμε στην ανταλλαγή απόψεων. Ο κύριος Έρνες Κούρτασουν, ο εισηγητής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τις τρεις ομιλήτριες για τις ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Κάποιες ερωτήσεις από την πλευρά μου. Κάποια στοιχεία πρέπει να τα εξετάσουμε. Είναι σαφές νομίζω ότι η πηγή ανισοτήτων λόγω φορολόγησης είναι μεγάλη. Μία ερώτηση πρώτα στην κυρία Κλάτσερ για τις συστάσεις αναχώρα και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Αυτό το πιέσαμε, το σπρώξαμε πολύ από την Επιτροπή μας. Όχι να έχουμε γενικές συστάσεις, αλλά να έχουμε και αξιολόγηση που άλλων ε, συστάσεων προκειμένου περί ισότητας. Τώρα, κάποιες συστάσεις ε, είπατε ότι είναι επικίνδυνες από την άποψη του φίλου. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν ε, προσθέθηκε μια σύσταση. Ποιες είναι αυτές που είναι επικίνδυνες, γιατί πρέπει να το εξετάσουμε αυτό. Να δούμε δηλαδή ποιες συστάσεις ε, υπονομεύουν την ισότητα των φίλων; Το άλλο ενδιαφέρον είναι το σχόλιο σας για την ε, περιβαλλοντική φορολόγηση. Είπατε ότι καμιά φορά δεν είναι ουδέτερη από άποψη φύλου. Διαισθητικά θα έλεγα ότι όταν ε, προχωρήσαμε στην οικολογική φορολογία θέλαμε να μειώσουμε τις επιβλαβείς για το περιβάλλον δραστηριότητες. Άρα θα ήταν η φορολογία αυτή ε, ουδέτερη από άποψη ή θα προωθούσε την ισότητα των φύλων. Εσείς όμως έχετε διαφορετική άποψη. Πρέπει να το δούμε αυτό γιατί είναι σημαντικό. Η τελευταία πρότασή σας για ένα συμβούλιο για την ισότητα και τα φορολογικά θέματα, αυτή η πρόταση είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν ξέρω αν προτείνεται να γίνει αυτό σε επίπεδο κρατών μελών, δηλαδή ένα σε κάθε κράτος μέλος, ή να έχουμε ένα μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν ισχύει το πρώτο, οι ανεξάρτητες φορολογικές αρχές δεν ξέρω αν θα μπορούσαν να βοηθήσουν, γιατί τώρα έχουμε διαφορετικές ανεξάρτητες φορολογικές αρχές και μπορεί να έχουν και κάποιες μονάδες για το φύλλο. Πάντως η πρόταση είναι ενδιαφέρουσα. Και τελευταία ερώτηση στην κυρία Γκούναρσον. Ε, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα που είπατε, βέβαια ε, ε, υπάρχει αυτή η συζήτηση γύρω από τον Πικέτη και την αλλαγή από τη φορολογία εργασίας στην φορολογία κεφαλαίου και είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε τον αντίκτυπο στα φύλλα, γιατί οι γυναίκες στηρίζονται περισσότερο στο εισόδημα εργασίας. Οπότε έτσι θα αυξάνονταν η ισότητα. Εσείς όμως έχετε στατιστικά στοιχεία που να δείχνουν ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι ε, τα έσοδα από κεφάλαια ε, αφορούν περισσότερο τους άνδρες. Κυρία Χάνη Παρασκιώδης. Ευχαριστώ πολύ τους ομιλητές. Ευχαριστώ και την Κομισιόν για το έγγραφο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο θέμα βέβαια. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα ξέρετε ότι τώρα μπήκε σε προεκλογική περίοδο και ως επιτοπλίστων όταν έχουμε προεκλογική περίοδο ε, συζητούμε τα φορολογικά. Πολύ. Τα περισσότερα από αυτά που είπατε δεν συζητούνται σε πολιτικές συζητήσεις για τη φορολόγηση, ενώ θα έπρεπε. Έχουμε διαφορετικούς φορολογικούς συντελεστές. Ε, ε, θα, πρέπει να δούμε αν η κυβέρνηση μπορεί να αυξήσει οδήματος, ΦΠΑ κλπ. Αυτά τα συζητούμε, αλλά δεν συζητούμε πώς είναι δομημένο ολόκληρο το φορολογικό σύστημα, ούτε εξετάζουμε τη διάσταση του φύλου. Οπότε ήταν πολύ καλά αυτά που μας είπατε για να αποκτήσουμε μια ιδέα του που βρίσκονται τα προβλήματα. Οι περισσότεροι μας γνωρίζουμε, θεωρώ, ότι ο ΦΠΑ, ο φορός κατανάλωσης και άλλοι είναι αντίστροφα προοδευτικοί και επιβαρύνουν τις γυναίκες. Και στο Ηνωμένο Βασίλειο οι φόροι εισοδήματος είναι πιο προοδευτικοί αλλά υπάρχουν και όρια στη λειτουργία του συστήματος και είναι λιγότερο προοδευτική ε, σε κάποια κράτη. Ε, είναι πολλά ενδιαφέροντα τα ε, θέματα εδώ. Και βέβαια το φορολογικό σύστημα έχει μια ενσωματωμένη διάκριση ανισότητας γιατί πολλές φορές το φορολογικό σύστημα αναπτύχθηκε αγνοώντας τα θέματα του φύλου. Ίσως λοιπόν θα έπρεπε να δουλέψουν περισσότερο οι γυναίκες στα θέματα φορολόγησης για να δουν μέσα από το δικό τους πρίσμα το θέμα αυτό. Αυτό δεν συμβαίνει συχνά. Υπάρχουν ορισμένα πραγματικά θέματα διάστασης του φύλου και διάρθρωσης του φορολογικού συστήματος και λειτουργίας του. Και πολύ σημαντικά είναι και όλα αυτά που είπατε για, την, ε, ε, τα καθήκοντα μέσα στην οικογένεια, γονικές άδειες, ε, άδεια μητρότητας, πατρότητας, αμοιβή. Και δείξατε ότι όλα αυτά επίσης έχουν αντίκτυπο. Επίσης σε γυράσκοντα πληθυσμό, ε, στους ηλικιωμένους, επίσης ε, υπάρχει αντίχτυπος γιατί οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής ε, κατά μέσον όρο. Καλό θα ήταν στην Επιτροπή μας λοιπόν να εστιάσουμε περισσότερο σε κάποια από αυτά τα θέματα. Έχουμε περιθώριο να κάνουμε πολλή δουλειά εδώ. Ευχαριστώ κύριος Γκέρκερ. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Κάναμε ένα άλμα στο, στην ισότητα. Ελπίζω να μ' ακούνε όλοι με τα ακουστικά. Ε, λοιπόν, κάποιες σκέψεις να εκφράσω. Όταν μιλάμε για φορολόγηση φιλική προς την ανάπτυξη, τι εννοούμε με growth, μεγέθυνση, ανάπτυξη. Από ό,τι γνωρίζω, στη Γαλλία από το τρίτο παιδί, μετά το τρίτο παιδί, δεν, πληρώνει κανείς, ε, δεν πρέπει να πληρώνει κανείς ε, φόρο εισοδήματος. Είναι αυτό η φορολόγηση φιλική προς την ανάπτυξη, δεν ξέρω. Τώρα, επίσης, ε, ανεξάρτητα από τις ελαφρύνσεις που θα πάρουν οι ηλικιωμένοι φορολογικά, αν πάρουμε το φόρο ΦΠΑ, μέσω των παιδιών τους πληρώνουν περισσότερα ως μη έχοντες παιδιά, που αυτό σημαίνει ότι ε, ε, ε, εξανεμίζονται οποιασδήποτε ελαφρύνσεις και βγαίνουν ζημιωμένοι στο τέλος. Κύριε Βαντάμ, προχωρήσατε πάρα πολύ μακριά με τη σκέψη σας. Το unpaid work, μια αμοιβόμενη εργασία. Εδώ θα ήθελα να δω τη διαφορά μεταξύ αυτών που έχουν παιδιά και των άτεκνων. Μιλάμε εδώ για παιδιά, όχι για παιδιά που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά, αλλά για την ε, σύγκριση της, ε, σε θέματα ισότητας. Πόση περισσότερη δουλειά έχουν οι γονείς από ότι οι άτεκνοι. Να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης εδώ. Ε, επίσης, όταν μιλάμε για την Parental Leave Directive, την οδηγία για τη γονική άδεια, Νομίζω ότι είμαστε πολύ χαμηλά σε σχέση με τους μήνες που προβλέπουμε. Μιλάτε για το Βέλγιο και τα 700 ευρώ. Εμείς όμως έχουμε 28 κράτη-μέλη και θα είναι δύσκολο να μεταφερθεί και αλλού το σύστημα αυτό. Ξέρετε πόσο στοιχίζει να πάει ένα παιδί σε ένα βρεφονιπιακό σταθμό ή σε ένα νηπιαγωγείο ε, τι σημαίνει αυτό ε, με μορφή ε, μισθού και πώς μπορεί να μεταφερθεί σε γονείς που φροντίζουν τα παιδιά στο σπίτι. Έτσι μπορούμε να έχουμε συγκρίσιμα μεγέθη. Και νομίζω ότι αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς της ισότητας. Όταν μιλάμε για χρηματοδότηση, στο Βέλγιο ποιος πληρώνει το, τη σύνταξη πληρώνουν οι επόμενες γενναίες ή ο καθένας ε, χρηματοδοτεί τη σύνταξή του. Αν γίνεται το πρώτο, αν πληρώνουν οι επόμενες γενναίες, τότε θα έλεγα τους άτεκνους που έχουν σημαντικά υψηλότερη σύνταξη, ε, αυτή η σύνταξη χρηματοδοτείται από τα παιδιά ξένων ανθρώπων. Και οι άτεκνοι εν προκειμένου Ε, θα μπορούσαν ε, συμμετέχουν στην χρηματοδότηση των επόμενων γενεών. Οπότε οι επόμενες γενναίες ε, δεν θα μπορούσαν να τα καλύψουν αυτά με μερική απασχόληση, για παράδειγμα. Αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα, αλλά μπορούμε να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. Και η κυρία Γκούναρσον μας είπε πολλά σημαντικά Είναι πολύ ωραία αυτά που μας είπατε. Και νομίζω ότι για τους γονείς ε, αυτό θα ήταν μια μεγάλη βοήθεια. Ευχαριστώ και εγώ για τις ομιλίες. Να προσθέσω κάτι ακόμα ε, που αφορά τη Γερμανία κυρίως. Στη Γερμανία, στα πλαίσια μιας συμβασίση, ε, υπάρχουν ε, κονδύλια που δίνονται στην Καθολική Ευαγγελική Εκκλησία. Αυτά είναι χρήματα από την φορολογία που ε, πληρώνουν οι πολίτες. Η υψηλή μισθή στην Εκκλησία πληρώνονται από το κράτος. Αυτή είναι μια ιδιαιτερότητα που δεν είναι γνωστή ευρέως. Δεν θέλω να το επικρίνω, εδώ και 200 χρόνια υπάρχει το σύστημα αυτό. Θέλω όμως να πω ότι εδώ υπάρχει σαφής αναδιανομή όλων των ε, φόρων που εισπράττονται στους άνδρες. Αφού στην Καθολική Εκκλησία όλοι οι ερωμένοι είναι άνδρες και οι επίσκοποι και όλοι. Ε, υπάρχει λοιπόν αυτή η συμφωνία ε, με τη μορφή νομικής βάσης που αφορά την αναδιανομή των φόρων που δεν είναι φόροι της που πληρώνει η Εκκλησία αλλά οι πολίτες. Και ε, αυτή είναι μια αναδιανομή που ζημιώνει τις γυναίκες και ε, εξυπηρετεί τους άντρες. Εκατο, πρόκειται για ε, 190 εκατομμύρια το χρόνο. Για λόγους ε, ισότητας ε, θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Αν έχουμε ε, ένα επάγγελμα, γιατί και το επισκόπου είναι ένα λειτουργήμα έστω, αλλά ε, μια επαγγελματική δραστηριότητα. Ε, αφού πρόκειται μόνο για άνδρες στην Καθολική Εκκλησία δεν μπορεί να χρηματοδοτείται από το, τα φορολογικά έσοδα του κράτους γιατί έτσι αποκλίνονται οι γυναίκες θα πρέπει να τονίσουμε ότι αυτό δεν είναι δίκαιο Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, οι ειδικοί να απαντήσουν, να αντιδράσουν στα σχόλια και στις παρατηρήσεις που ακούστηκαν. Δύο λεπτό καθένας όμως μόνο έχετε, γιατί πρέπει να ψηφίσουμε σε νέα λεπτά. Δύο λεπτό καθένας λοιπόν για τις απαντήσεις. Παρακαλώ. Δύο λεπτά για τόσο πολλές ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω. Καταρχήν, οι συστάσεις. Για παράδειγμα, για τον περιορισμό της χρήσης των περιορισμένων ποσοστών ΦΠΑ. Αν ξέρουμε ότι η ΦΠΑ μειώνεται, τότε το βάρος το απομονίζονται περισσότερο οι γυναίκες. Για το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματο θα πηγαίνει είναι κάτι επικίνδυνο. Η πρόταση για την μείωση του εταιρικού φόρου επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη βάσει της κατανομής. Είναι πράγματα κάπως επικίνδυνα. Και γι' αυτό πρέπει κάθε φορά να γίνονται εξελογήσει αντικτύπου πριν από οποιαδήποτε απόφαση. Δεύτερον, για την περιβαλλοντική φορολογία και πάλι εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες. Ας δούμε ε, το φόρο του διοξιδίου του άνθρακα. Αν επιβληθεί στη βενζίνη, το ενεργειακό κόστος μπορεί να αυξηθεί. Και τότε ε, επιβαρύνονται περισσότερο τα χαμηλότερα εισοδήματα. Άρα οι γυναίκες. Γιατί δυστυχώς ακόμα σε όλες μας τις χώρες εκείνες είναι στα χαμηλότερα εισοδήματα αλλά υπάρχουν και άλλες πτυχές. Γιατί υπάρχουν πολιτικές άμβλησης και πώς υλοποιούνται, πώς εφαρμόζονται. Τι γίνεται επίσης με τα φορολογικά έσοδα από τον περιβαλλοντικό φόρο. Θέλω δηλαδή να τονίσω ότι οποιοδήποτε φορολογικό φόρος, έτσι κι αλλιώ έχει επιπτώσεις επί της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων. Και φυσικά είναι κάτι πολύ σημαντικό, αλλά θα πρέπει να ελεγχθεί προηγουμένω πολύ καλά ποιο είναι ο αντίκτυπο. Καλό θα ήταν να έχουμε ένα καλό πλαίσιο για την ανάλυση, να αναλύσουμε πρώτα απ' όλα τι ήδη υπάρχει Υπάρχουν μελέτες και κάποιες από αυτές έχουν ένα καλό πλαίσιο, λαμβάνουν υπόψη δηλαδή τη σχέση αυτή με την ισότητα. Λέμε ότι ο φόρος πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε να ενισχύεται η ανάπτυξη. Το πρόβλημα εδώ είναι Πρώτον, ότι οι περικοπές στους φόρους δεν είναι σίγουρο ότι οδηγούν εκεί για το οποίο προβλέθηκαν και έπειτα υπάρχει ένα μεγάλο κόστος λόγω των ε, μεγάλων διαφορών που απορρέουν από την φορολογική πολιτική. Και όσον αφορά την ε, ισότητα και την φορολογική συμπεριφορά και τα φορολογικά συμβούλια, θα πρέπει να γίνεται κάτι και σε επίπεδο χωρών μελών και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά προτείνω οι αρχές να είναι χωριστές. Γιατί αν ε, είναι ενιαία, τότε οι άνθρωποι εκεί θα ασχολούνται ε, με μερική απασχόληση και κάπου θα χάνονται όλα αυτά. Είναι καλύτερα να πούμε ότι χρειαζόμαστε συμβούλια εμπειρογνωμόνων ειδικά για την ισότητα και τη φορολογική πολιτική και όχι να είναι γενικώ κάποια συμβούλια ισότητα για τα πάντα. Ευχαριστώ κύριο Βαντάμε. Ευχαριστώ και εγώ και ευχαριστώ για τις ερωτήσεις και τον κύριο Γκέρικε. Εγώ δεν είμαι τόσο συνηθισμένος στην ταυτόχρονη μετάφραση, λέει ο μιλητής, οπότε δεν είμαι σίγουρος αν σας κατάλαβα κατάλαβα πολύ καλά για αυτά που είπατε, για τα κίνητρα ε, υπέρ των αντρών, όχι, ώστε οι άντρες να υποφελούνται περισσότερο από τη γονική άδεια. Δεν ήταν αυτό που είπατε. Ναι, αφενός μεν. Αν υπάρχουν ε, όντως αμοιβέ που προβλέπονται, οι άντρες θα το κάνουν, αλλά δεν θέλουν φιλοδόρημα. Αυτό θέλω να πω. Αν περάσουμε από τους τέσσερις μήνες με 700 ευρώ το μήνα, που δεν είναι τόσο ελκυστικό γιατί όντως χάνει κανείς έσοδα, και πάμε στους δυόμισι μήνες με 1.500 ευρώ το μήνα, που είναι κάτι παραπάνω από το μέσο μισθό στο Βέλγιο στο κάτω-κάτω, τότε νομίζω ότι αντισταθμίζεται η απώλεια εισοδήματος και έτσι δίνονται κίνητρα στους άντρες να παραμείνουν στο σπίτι μετά τη γέννηση του παιδιού τους. Βέβαια, σε έναν ιδανικό κόσμο θα ήταν ακόμα περισσότερο και μου αρέσει το σουηδικό σύστημα όπου τα ζευγάρια έχουν και ένα μπόνους εφόσον μοιραστούν εξίσου τη γονική άδεια μετά τη γέννηση του παιδιού τους. Θα μπορούσαμε να πάμε ακόμα πιο μακριά. Αλλά η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας μου δεν είναι τόσο λαμπρή όπως εκείνη της Σουηδίας ή της Νορβηγίας, δυστυχώς. Τώρα για τη δεύτερη ερώτησή σας είπατε ότι αυτό το επιπλέον κόστος σε ένα σύστημα κατανομής επιβαρύνει τις νέες γενιές, έτσι, τους νέους. Η ερώτησή μου ήταν ότι εάν χρηματοδοτούνται οι συντάξεις από τις επόμενες γενιές, τότε πρέπει να αναρωτηθούμε ποιος χρηματοδοτεί τις επόμενες γενιές. Και δεν είναι ευθύνη μόνο των γονιών να πληρώνουν, αλλά να πληρώνουν και αυτοί που δεν έχουν παιδιά για να χρηματοδοτήσουν αυτές τις συντάξεις. Με φόρους που θα πηγαίνουν ε, στις συντάξεις, για παράδειγμα. Απάντηση. Φυσικά και υπάρχει φοροπαλλαγή. Πληρώνουν λιγότερους φόρους οι γονείς, δηλαδή τα ζευγάρια χωρίς παιδιά πληρώνουν περισσότερου φόρου. άρα συνεισφέρουμε με αυτόν τον τρόπο. Έπειτα το λεγόμενο marital quotient, αν δείτε την αναλογία ή τα ωφέλη, Η μεταρρύθμιση αυτής της αναλογίας σημαίνει ότι πηγαίνει ποσοστό από τις ε, παλιότερες γενιές στις νέες γενιές. Παρακαλώ και εσείς τώρα. Εκτός μικροφώνου ομιλήτρια, δεν την ακούμε. Ναι, φυσικά και υπάρχουν στατιστικά δεδομένα και θα μπορούσαμε να συγκεντρώσουμε κι άλλα. Πάντως, είναι γνωστό ότι όταν πρόκειται για οικονομικά μέσα, οι γυναίκες είναι απούσες είναι παρούσες όταν μιλάμε για αποταμίευση, για οικονομίες. Αλλά έχουμε αρνητικά έτσι κι αλλιώς ε, επιτόκια. Οπότε η οικονομική ανάπτυξη ή εν πάση περιπτώσει όταν πρόκειται για τις κεφαλαγορές και τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, τότε έχουμε μεγαλύτερη απόδοση και εκεί έχουμε μόνο τους άντρες. Υπάρχουν μελέτες συμπεριφορά και τα λοιπά. Γιατί οι γυναίκες δεν αναλαμβάνουν τέτοιους κινδύνους στις κεφαλαιαγορές, να το συζητήσουμε. Αλλά περί αυτού πρόκειται και επανερχόμαστε στο βασικό θέμα. Αυτή η κοινωνική νοτροπία που υπάρχει και διαφοροποιεί άντρες και γυναίκες. Έχουμε φτάσει σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον ζήτημα για το πώς οι καθολικοί ιερείς πληρώνονται από το φορολογικό σύστημα, από τη φορολογία, τα φορολογικά έσοδα. Πολλοί Γερμανοί μπορεί να πιστεύουν ότι είναι ουδέτερο. Και σε άλλες χώρες μέλη μπορεί να υπάρχουν αντίστοιχες ε, φορολογικές πρακτικές. Ρυθμίσεις που θεωρούνται εντελώ ουδέτερες, εντελώ κανονικές και φυσιολογικές, αλλά τελικά δημιουργούν αυτήν την διαφορά μεταξύ των δύο φύλων. Βεβαίως, μέσω του φορολογικού είμαστε έτοιμοι να πληρώσουμε για ένα ακριβό σύστημα ε, φορολογικό στη Γερμανία ή στη Γαλλία. Κοστίζουν πολύ Νομίζουμε ότι αξίζει τον κόπο όμως, δεν τον φυσβητούμε. Και όταν φτάνουμε σε μια μεταρρύθμιση για τη γονική άδεια, τότε αρχίζουν οι συζητήσεις πώς θα χρηματοδοτηθεί. Βλέπετε δηλαδή ότι υπάρχει διαφορά στην αντιμετώπιση του φορολογικού που δεν είναι στα χέρια των γυναικών. Και ερχόμαστε σε αυτό που λέει και η κυρία Χάνιμπολ. Ναι, χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα να γίνουν για τη συνειδητοποίηση των ε, διαφορών και των δυνατήτων που υπάρχουν για την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Βοηθήστε μας, είσαστε ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και εσείς η δική σας επιτροπή, εσείς έχετε την εξουσία να το κάνετε, δεν την έχω εγώ. Εγώ είμαι πολύ μόνη όταν πρόκειται για τέτοια ζητήματα. Εσείς μπορείτε να συνεισφέρετε. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους ομιλητές, τους ειδικού μας και όλους τους ευρωβουλευτές που συμμετείχαν σε αυτή τη συζήτηση. Όντως οι πληροφορίες που πήραμε ήταν πολύτιμες και θα μας βοηθήσουν να προετοιμάσουμε την έκθεση Δίας Πρωτοβουλίας που θα έχουμε σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν όλους. Θα αρχίσουμε την ψηφοφορία σε κάνα δύο λεπτά. Ετοιμαστείτε παρακαλώ.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 Λοιπόν, συνάδελφοι, είστε έτοιμοι για την ψηφοφορία. Προφορική ερώτηση. Τερματισμός των γάμων των παιδιών. Ε, πρώτο κομμάτι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Τελική ψηφοφορία στο κείμενο όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Επόμενο για τη διάσταση του φύλου Ε, διεθνές εμπόριο και εμπορικές πολιτικές στη παγκόσμια διαρξιακή αλυσίδα. Η τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 10. Προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Και σε χωριστή ψηφοφορία, πρώτο τμήμα σε τμήματα, κατά, αποχές δεκτό και δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτό. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Έλεγχος, έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 13. Σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Δεύτερο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά θα ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτό. Με διαφορά μιας ψήφου. Τροπολογία 14. Σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος. Πέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές, δεκτό. Τροπολογία 15 σε δύο τμήματα. Πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Τροπολογία 16 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Αιτιολογικές σκέψεις. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχει σήμερα άλλες ψηφοφορίες. Και Προχωρούμε στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης. will uh, Συνεχίζουμε, συνάδελφοι. Σημείο 8. Ανάγκη για ενωσιακή στρατηγική που θα θέσει τέλος και θα προλάβει το συνταξιοδοτικό κενό μεταξύ των φίλων. Ε, θα δώσω το λόγο στην κυρία Ανιέσκα Κλόν Ντόμιντσάκ από την Οικονομική Σχολή της Βαρσοβίας. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσω την έκθεση αυτή για τις διαφορές στις ε, συντάξεις, όχι τις σημερινές, αλλά εξετάζουμε τις δυνατότητες για τη μείωση της διαφοράς, λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή κατάσταση των γυναικών στην αγορά εργασίας γιατί είναι χρήσιμο να προσπαθήσουμε να το δούμε αυτό προοπτικά. Αυτό το οποίο βλέπουμε στην παρούσα φάση έχουμε να κάνουμε με συστήματα τα οποία έχουν σχεδιαστεί στο παρελθόν. Υπάρχουν όμως πολλές αλλαγές στον τρόπο απασχόλησης των γυναικών, το είδαμε αυτό τα τελευταία χρόνια η γύρανση του πληθυσμού έχει οδηγήσει σε αναθεωρήσεις των συνταξιοδοτικών συστημάτων, αύξηση του χρόνου απασχόλησης και εισαγωγή μια μικρή. Look like in the future. Uh, women participation on the labor market also changes. In some countries, women work longer because of higher retirement ages or because of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 ο οποίος ε, επεκτείνει την ανάλυση των κενών αυτών πέρα από μεμονωμένους δείκτες που θα λαμβάνονται υπόψη σε σχέση δηλαδή με μισθούς, απασχόληση ή επίπεδα σύνταξης, θα δώσει μια προοπτική σε σχέση με τον αντίκτυπο των συνδυασμό διαφορετικών παραγόντων που συμβάλλουν στις διαφορές φύλους στις συντάξεις, όχι μόνο τώρα αλλά και στο μέλλον. Και ενθαρρύνει και θα ήθελα και εμείς να συζητήσουμε θέματα όπως γιατί κάποιες χώρες ε, ε, έχουν καλύτερα αποτελέσματα από ότι άλλες. Ή το σχεδιασμό των συνταξιδοτικών συστημάτων πώς επηρεάζει αυτά τα κενά μεταξύ φύλων. τι σημαντικό, πώς αλληλεπιδράει η το σχεδιασμο των συνταξιοδοτικων συστηματων πως επηρεαζει αυτα τα κενα μεταξυ εργασίας στα συστήματα συνταξιοδότηση σε σχέση με το κενό μεταξύ, και το χάσμα μεταξύ ε, γενεών. Ε, πολλές φορές όλα αυτά είναι αποτέλεσμα του τι συμβαίνει κατά το χρόνο εργασίας. Ε, δηλαδή πόσο συμμετέχουν οι γυναίκες στην αγορά εργασίας, τι ύψος μισθού έχουν κλπ. Για να υπολογίσει κανείς ε, το κενό αυτό πρέπει να προσπαθήσει να βρει μία λύση η οποία να βασίζεται σε ορισμένες αρχές και ορισμένα χαρακτηριστικά. Βασικό είναι η συγκρισιμότητα ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να υπολογίσουμε τα επίπεδα των συντάξεων στο μέλλον για τις γυναίκες και τους άνδρες θα πρέπει να βασίζεται σε δείκτες οι οποίοι να είναι συγκρίσιμοι μεταξύ τους, ενοποιημένοι στατιστικά ή ε, όμοιοι στατιστικά. Θα πρέπει να είναι επίσης ε, βιώσιμοι οι δείκτες αυτοί. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπολογίζονται σε τακτική βάση και γι' αυτό προτείνουμε τον συγκεκριμένο δείκτη. Θα πρέπει επίσης να έχουν ένα αυστηρά υπολογισμένο αποτέλεσμα το οποίο να λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό των συντάξεων. Θα πρέπει να βασίζεται στην τρέχουσα γενεά εργαζομένων γυναικών, γιατί αυτή τη στιγμή πληρωθούν οι συντάξεις. Υπάρχουν πάρα πολύ λίγα τα οποία μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξουμε το επίπεδο των συντάξεων αυτών αλλά οι πολιτικές μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο θα σωρευτούν ε, τα νέα ένεργα για τον υπολογισμό των επιπέδων σύνταξης. Και τέλος είναι το θέμα της κάλυψης. Ο τρόπος με τον οποίο προτείνουμε, καλύπτουμε όλες τις χώρες, 28 χώρες, και επίσης και για χώρες πέραν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να έχουμε πληρέστερες συγκρίσεις. Τώρα πόσο δημιουργείται ο συγκεκριμένος δείκτης. Όπως σας είπα έχουμε δύο τομείς. Ο ένας έχει σχέση με το συνταξιοδοτικό σύστημα και ο άλλος με την εργασία. Ο κλάδος της εργασίας καλύπτει το 65% των στοιχείων. Αυτό οφείλεται στο ότι οι περισσότερες από τις διαφορές στα επίπεδα των συντάξεων συμβαίνουν λόγω ακριβώς των διαφορών στην ίδια την αγορά εργασίας. Πρόκειται για μια πρόταση υπολογισμού της συγκεκριμένης αυτής διαφοράς και εμείς στην Πολωνία αναλύσαμε τον τρόπο με τον οποίο δίδονται οι ελάχιστες, οι χαμηλότερες συντάξεις και είδαμε ότι η διαφορά ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες οφείλεται απλά στους χαμηλότερους μισθούς των γυναικών κατά τη διάρκεια της ε, εργασιακής τους δραστηριότητας. Οι δείκτες τώρα, οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη στον τομέα της απασχόλησης, είναι πρώτον ο χρόνος εργασίας, αν υπάρχει διαφορά, ε, με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουμε για την απασχόληση σήμερα των γυναικών, συγκρίνουμε το τι συμβαίνει σήμερα με το τι συνέβαινε πριν από 40 χρόνια. Αυτό είναι θα έλεγα μια διάρκεια γενεάς η οποία λαμβάνεται υπόψη. Κάνουμε μια προβολή των στοιχείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των στοιχείων των κρατών μελών λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εργαζόμενος ο μέσος δουλεύει γύρω στα 30 χρόνια. Είναι ένας δείκτης αυτός, ο θεωρητικός εν πολλής. Ο δεύτερος δείκτης είναι η διαφορά στις αμοιβέ και ο τρίτος είναι η διαφορά στην ένταση της εργασίας. Ε, γιατί εδώ λαμβάνουμε υπόψη τις γυναίκες οι οποίες έχουν μερική απασχόληση, δεν έχουν πλήρης απασχολήσει. Ε, δεν έχουν πλήρης αμοιβέ, έχουν χαμηλότερες συντάξεις. Τώρα, στη δεύτερη πλευρά, στο 35% στο σύστημα των συντάξεων, ε, καταρχάς επανέρχομαι στην απασχόληση να πω ότι λαμβάνουμε υπόψη και τις μεταβλητές οι οποίες χαρακτηρίζουν τα ποσοστά απασχόλησης και επίσης και τα συστήματα αναπλήρωσης και έρχομαι τώρα στο σύστημα το συνταξιοδοτικό. Οι μελέτες που έχουμε εδώ και λίγα χρόνια μας δείχνουν ότι μπορούμε να έχουμε μία προοπτική για τα επόμενα τρία χρόνια μόνο. Καταρχάς αντιστάθμιση για διακοπή επαγγελματικής δραστηριότητας. Μια γυναίκα η οποία σπάει την καριέρα της για τρία χρόνια για να γεννήσει και να μεγαλώσει το παιδί τι συνέπειες έχει αυτό. Δεύτερον, η αναδιανομή των συνταξιοδοτικών αμοιβών στην ουσία είναι ε, η σχέση ανάμεσα στο θεωρητικό επίπεδο αναπλήρωσης του εργαζομένου, ο οποίος παίρνει τα δύο τρίτα του μέσου μισθού κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, επειδή ακριβώς οι γυναίκες έχουν χαμηλότερη διάρκεια απασχόλησης, ωφελούνται από την ανακατανομή της συνταξιοδοτική θεωρητικά. Ταυτόχρονα, ο δείκτης ε, της ε, σύνδεσης ε, της σύνταξης λοιπόν που δίδεται με την προβλεπόμενη τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ βλέπουμε ότι οι γυναίκες θεωρητικά εφόσον εργαστούν περισσότερο από τις ζουν περισσότερο από τους άνδρες και γι' αυτό θεωρητικά θα πάρουν συντάξεις για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Και το τελευταίο κομμάτι του δίκτυα αυτού είναι η διαφορά στα επίπεδα της ε, συνταξιοδότησης λόγω ηλικίας. Σε πάρα πολλές χώρες είναι περίπου ίδιο το ανώτατο όριο, αλλά μερικές φορές υπάρχουν διαφορές όπως Σλοβενία, Πολωνία, Ρουμανία και Βουλγαρία. Στις τέσσερις αυτές τις χώρες υπάρχουν διαφορές μεγαλύτερες από τις όλες προηγούμενες. Ο χάρτης εδώ δείχνει ε, τον υπολογισμό της διαφοράς ε, Τσεχία, Φιλανδία, Σουηδία και τα λοιπά είναι χώρες οι οποίες έχουν το χαμηλότερο ποσοστό, έχουν ε, ικανοποιητική συμμετοχή των γυναικών στην εργασία, έχουν χαμηλότερα ποσοστά μερικής απασχόλησης και παρόμοια επίπεδα συντάξεων. Ενώ υπάρχουν χώρες όπως η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Ελλάδα και η Ιταλία έχουν πολύ μεγάλες διαφορές στις συντάξεις διότι οι γυναίκες έχουν πολύ χαμηλότερες αμοιβέ και ταυτόχρονα στην Ολλανδία έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών που εργάζονται part-time σε μερική απασχόληση και αυτό επηρεάζει και δίνει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις συντάξεις. Λοιπόν, συμπερασματικά τώρα ότι οι χώρες οι οποίες έχουν υψηλό δίκτυ, έχουν υψηλή απασχόληση του στις γυναίκες που εργάζονται πλήρως, συνήθως έχουν αντιστάθμιση και αποζημίωση για τη διακοπή της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, έχουν αναδιανομή των συστημάτων των συνταξιοδοτικών προς τους χαμηλά αμοιβόμενους. Θα ήθελα να πω επίσης να πω κάτι για την διαφορά στην γυναική απασχόληση ανάμεσα στις διάφορες χώρες, κάτι το οποίο δίδει πολλές εξηγήσει για τη σημερινή κατάσταση. Εδώ βλέπετε την κατανομή των ποσοστών απασχόλησης ηλικιακά και δείχνει τις υψηλότερες αξίες και τις χαμηλότερες αξίες στις χώρες της Ένωσης. Η πράσινη γραμμή είναι ο μέσος όρος και βλέπετε κάτω και πάνω της άνω τα δύο άκρα. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη και οι διαφορές αυτές είναι πάρα πολύ σημαντικές στις χώρες με υψηλές συντάξεις. Σε ορισμένες χώρες υπάρχουν δυνατότητες για πρόορη συνταξιοδότηση των γυναικών, σε άλλες όχι. Και φυσικά όσο λιγότερο εργάζεται κάποιος, τόσο χαμηλότερο είναι και το επίπεδο της σύνταξης, σύνταξης την οποία θα πάρει. Αν δούμε τώρα την διαφορά που ισχύει σήμερα στις συντάξεις επί τη βάση των αξιών τις οποίες μας, ε, των στοιχείων τα οποία έχουμε ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες, βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες θετικές εξελίξεις, υπάρχουν όμως και χώρες οι οποίες πηγαίνουν αρκετά καλά, έχουν καλά αποτελέσματα και δεν θα έχουν να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα μεγάλου κενού, μεγάλης διαφοράς στο μέλλον λόγω της εξέλιξης των συνταξιοδοτικών συστημάτων. Κάποια συμπεράσματα λοιπόν. Θα πρέπει να ενισχύσουμε πολιτικές που έχουν σαν στόχο τη μείωση των διαφορών στην αγορά εργασίας ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες. Να διευκολύνουμε την πρόσβαση από την κατάρτιση και τη σχολική εκπαίδευση στην εργασία όπου οι γυναίκες έχουν πολύ υψηλότερους κινδύνους να μείνουν εκτός της επαγγελματικής κατάρτισης και γι' αυτό χρειάζονται στήριξη, κάτι το οποίο μπορεί να επηρεάσει τις δυνατότητες που θα έχουν στην αγορά εργασίας. Πρέπει να ενισχύσουμε την δυνατότητα συνδυασμού και συμφιλίωσης της εργασίας και της οικογένειας, και να έχουμε υψηλά επίπεδα προστασίας και υποδοχής ε, παιδιών και ε, φροντίδας γενικότερα. Θα πρέπει να υπάρξει επίσης ε, κίνητρο για την επέκταση, την παράταση θα έλεγα της εργασιακής δραστηριότητας, κάτι το οποίο έχει υπογραμμιστεί συχνά. Υπάρχουν και κάποια, κάποια συμπεράσματα το αναδιανεμητικό σύστημα δεν μπορεί να αντικαταστήσει, ε, θα έλεγα, ένα ισότιμο σύστημα, αλλά θα πρέπει να παρακολουθούνται τα συστήματα αυτά για το πώς ε, family members για το πώς τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα θα κατανέμονται όχι μόνο σε σχέση και με τη φροντίδα των παιδιών αλλά και τη φροντίδα των υπολείπων μελών της οικογένειας θα πρέπει να υπάρξει εξίσωση των δυνατοτήτων συνταξιοδότησης ηλικιακών ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες και θα πρέπει επίσης να υπάρξουν και μέτρα που θα μειώσουν την διαφοροποίηση των επιπέδων συντάξεων ανάμεσα στις, ε, στους ηλικιωμένους άνδρες και γυναίκες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά τα ενδιαφέροντα που μας είπατε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχω ένα σχόλιο και μία ερώτηση, λέει η κυρία Κόσλαυσκα. Θέλω να ευχαριστήσω ε, την ε, εμπειρογνώμονα για αυτά που μας είπε. Πιστεύω ότι το θέμα αυτό του χάσματος είναι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που συζητάμε σε αυτή τη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και είμαστε μόνο στην αρχή τώρα που αναλύουμε το θέμα. Μας περιμένει πολλή δουλειά δηλαδή. Είναι η πρώτη ανάλυση που κάνουμε, είναι πολύ σημαντικός ο δείχτης αυτός για το μέλλον. Αυτό που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι εσείς αναφερθήκατε στις αιτίε και στον μηχανισμό της διαφοράς αυτής και αναφερθήκατε στο στοιχείο της αγοράς που έχει να κάνει δηλαδή με τη συμμετοχή των γυναικών ε, στην αγορά, πόσο έχουν δουλέψει, ε, part-time, μερική απασχόληση, πλήρη απασχόληση. Και υπάρχει και κάτι διαφορετικό που έχει να κάνει με την συνταξιοδότηση που είναι κάτι πιο ελκυστικό για τους πολιτικούς, γιατί για τους πολιτικούς είναι πιο εύκολο να αλλάξουν κάτι στο στοιχείο αυτό της συνταξιοδότησης αντί να κάνουν κάτι για την αγορά εργασίας. Και η έκθεσή σας δείχνει ότι το στοιχείο αυτό που έχει να κάνει με την αγορά, δηλαδή πόσα χρόνια δουλεύουν οι γυναίκες, είναι κάτι πολύ σημαντικό για τα δικαιώματά τους στα συνταξιοδοτικά. Πάνω σε αυτό λοιπόν πρέπει να επικεντρωθούμε και έρχομαι τώρα στις ερωτήσεις μου. Πρώτον, διαπίστωσα ότι σε ένα τμήμα της έκθεσης λέτε ότι οι μητέρες είναι περισσότερο θύματα του συστήματος. Κυρίως οι μητέρες που έχουν πάνω από δύο παιδιά, όσο πιο πολλά παιδιά έχουν δηλαδή, τόσο πιο πολλοί βουλιάζουν σε αυτό το πρόβλημα. Μπορείτε να πείτε κάτι περισσότερο γι' αυτό. Και η δεύτερη ερώτησή μου έχει να κάνει με τη μεθοδολογία. Γιατί είπατε ότι είναι δύσκολο να βρούμε συγκρίσιμα δεδομένα. Χρειαζόμαστε όμως δείκτες και εσείς προτείνετε έναν δείκτη που θα μας βοηθήσει να αξιολογήσουμε, να εκτιμήσουμε που βρισκόμαστε. Χρειαζόμαστε κάποιον δείκτη πρόβλεψης και να αξιολογήσουμε βάση αυτού του κριτηρίου. Όσον αφορά την μεθοδολογία λοιπόν υπάρχουν δεδομένα τα οποία θα μας βοηθούσαν να καταλήξουμε σε ένα τέτοιο δίκτυο ή άλλους ε, δείκτες και τι γίνεται με τα δεδομένα τα οποία δεν είναι συγκρίσιμα ή δεν υπάρχουν. Μπορούμε να τα βρούμε ή μπορούμε να κάνουμε μια προβολή, να τα υποθέσουμε ώστε να καταλήξουμε σε συγκρίσιμα δεδομένα. Και τι πρέπει να κάνουμε για να έχουμε καλά συγκρίσιμα στοιχεία, τα οποία θα μας επιτρέψουν να καταλήξουμε σε δείκτες, να φτιάξουμε δηλαδή δείκτες που θα μας βοηθήσουν στη συνέχεια. σε ευχαριστούμε. Δεν βλέπω άλλες ερωτήσεις, ούτε άλλο σχόλιο, οπότε παρακαλώ να απαντήσετε σε ερωτήσεις της κυρίας Κοσλόσκα. Ευχαριστώ πολύ. Απαντάει στα πολωνικά η ομιλία και συνεχίζει αγγλικά. Μάλλον συνεχίζει Υπάρχουν ε, διάφορα προγράμματα στην Ευρώπη και διάφοροι μηχανισμοί που αντισταθμίζουν τη διακοπή στη σταδιοδρομία. Υπάρχουν ε, κάποιες χώρες ε, που έχουν τις δικές τους λύσεις. Στη Γερμανία υπάρχει μια λύση όπου για κάθε παιδί οι γονείς έχουν κάποιο συνταξιδιωτικό μπόνους ανάλογα με το αν όντω διέκοψαν την ε, σταζιοδρομία του ή όχι. Δηλαδή μπορεί να καταλήξουν σε υψηλότερη σύνταξη από ότι τα ζευγάρια που δεν έχουν παιδιά. Ε, στην Πολωνία υπάρχουν διαφορετικές λύσεις για την γονική άδεια. Και οι δύο γονείς εφόσον πάρουν την γονική τους άδεια μπορεί να έχουν παραπάνω κατά 60%. Δηλαδή να κερδίσουν όσον αφορά την σύνταξή τους, αντί να έχουν μειωμένη σύνταξη επειδή διέκοψαν τη σταδιοδρομία τους. Η κάθε χώρα έχει τις δικές της λύσεις πάντως. Και εμείς αναφερόμαστε σε έναν δείκτη που μπορεί να βοηθήσει στην πρόβλεψη της αντιστάθμισης που χρειάζεται για αυτούς που διέκοψαν τη σταδιοδρομία τους σε σχέση με αυτούς που δεν την διέκοψαν. Άρα με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πούμε σε τι βαθμό τα καταφέρνουμε. Βέβαια, η κατάσταση είναι διαφορετική από χώρα σε χώρα. Οι χώρες που δίνουν μεγαλύτερη αντιστάθμιση για την διακοπή στη σταδιοδρομία θα έχουν και μικρότερες διαφορές στις συντάξει τελικά ανάμεσα στα δύο φύλλα. Είναι πολύ σημαντικός παράγοντας αυτός και σε μερικές περιπτώσεις όντως η σύνταξη μιας γυναίκας που διέκοψε τη σταδιοδρομία της για να μεγαλώσει τα παιδιά της έχει χαμηλότερη από εκείνη μιας γυναίκας που δεν διέκοψε επειδή έκανε παιδιά ακόμα και αν έχουν δουλέψει τον ίδιο αριθμό ετών. Συνήθως μιλάμε για τρία χρόνια. Αν όμως η διακοπή είναι πάνω από τρία χρόνια, θα έπρεπε να αναλύσουμε περισσότερο σε βάθος. Όσον αφορά πάντως τη μεθοδολογία, βασίζεται σε δείκτες που ίσως είναι συγκρίσιμοι σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρησιμοποιούμε δεδομένα πρώτα απ' όλα από την έρευνα για την αγορά εργασίας. Έπειτα χρησιμοποιούμε πληροφορίες οι οποίες αξιολογούνται βάσει της μελέτης μας για τις συντάξεις. Πρόκειται για κάτι σταθερό. Κάθε τρία χρόνια γίνεται αυτή η αξιολόγηση. Έχουμε λοιπόν τους δείκτες για το 2013. Επειδή το 2013 οι δείκτες αυτοί για τις συντάξεις αξιολογήθηκαν τότε και οι επόμενοι θα εκπονηθούν βάσει των στοιχείων που θα έχουμε για το 2016 και θα είναι έτοιμοι σε δύο χρόνια. Μπορούμε Πάντα βέβαια να έχουμε καλύτερες πληροφορίες. Η ιδανική κατάσταση θα ήταν να βασιζόμαστε σε υπάρχοντα δεδομένα για πολλά χρόνια και να οδηγηθούμε σε προσωμιώσεις και έτσι και σε προβλέψεις για τη συντάξη ανδρών και γυναικών. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια μέθοδος αρκετά περίπλοκη που χρειάζεται και αρκετό εργατικό δυναμικό. Δεν ξέρω αν όλες οι χώρες διαθέτουν κάτι τέτοιο. Πάντως ο δείκτη που προτείνεται τώρα είναι κάτι σαν ένα θερμόμετρο που μας βοηθάει να μετρήσουμε γενικά τον κίνδυνο που υπάρχει στο μέλλον να υπάρχουν διαφορές στις συντάξεις ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες. Πάντως, έχει να κάνει με την εργασία, με τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας. Κάποιοι συμμετέχουν 40 χρόνια και παραπάνω. Οπότε αν κάποιος συμμετέχει 40 χρόνια στην αγορά εργασίας, οι διαφορές συσσωρεύονται. Γιατί οι γυναίκες κερδίζουν λιγότερα. Η συσσόρευση αυτή οδηγεί σε μεγάλες διαφορές στη στιγμή της συνταξιοδότησης. Είναι ζωτική σημασία πάντω για το συνταξιδοτικό. Αν συγκρίνουμε το συνταξιδοτικό κεφάλαιο για τους άντρες και τις γυναίκες, ανεξάρτητα από την αντιστάθμιση, ο μηχανισμός αντιστάθμισης δεν τα καταφέρνει να καλύψει τις διαφορές που έχουν συσσωρευτεί για 40 χρόνια. Μπορούμε να κάνουμε κάποιες διορθώσεις, κάποιες προσαρμογές, αλλά οι επιπτώσεις υπάρχουν. Χρειάζεται λοιπόν ένα πραγματικό σύστημα αντιστάθμισης. Και πρέπει να προσέξουμε οι αντισταθμίσεις που γίνονται για το κάθε στάδιο, για την κάθε φάση, να μην οδηγήσουν σε αντίθετο αποτέλεσμα, σε μια υπερβολική αντιστάθμιση δηλαδή τη στιγμή της συνταξιοδότησης. Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση και για την απάντηση και τις στην ε, ερώτηση που σας έγινε από τη συνάδελφο. Ωραία. Αυτό ήταν το τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη, συνάδελφοι. Να σας υπενθυμίσω ότι η επόμενη συνεδρίαση θα είναι 8 Ιουνίου 9 το πρωί. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ και τους διερμηνήσε. Ευχαριστούμε πολύ.